Στις 21 Ιανουαρίου διακόπτει η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορούμε να συνεχίσουμε να επαναλάβουμε την Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα πρακτικά το...